Καλημέρα, συνάδελφοι. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ευρωεκλογές το 2014. Θα ήθελα να επενθυμίσω στους βουλευτές ότι για αυτή τη συζήτηση δεν προβλέπεται η διαδικασία του Catch the Δίνω το λόγο αμέσως στον Επίτροπο Σεμέτα. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντα πολύ σημαντικές στιγμές για την Ένωση και οι εκλογές του 2014 έρχονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα υποστήριζε κάθε προσπάθεια για την ενισχύση της νοημότητας του Κοινοβουλίου,